τα ορισμών της επιτροπές και τι αντιπροσωπείε. Αυτές οι, αυτοί ορισμοί θα υπάρχουν στα πρακτικά αυτή τη συνόδου. Αν δεν υπάρξουν δε παρατηρήσεις, μέχρι ότου να εγκριθούν τα, τα πρακτικά, οι διορισμοί αυτοί θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφάσισε να ξεκινήσει